Ας κάνουμε μία λοιπόν πρώτα δοκιμαστική ψηφοφορία. Έχετε βάλει όλες τις κάρτες σας να κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξεκινάει λοιπόν η ψηφοφορία. Πατήστε τα κουμπιά.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 Μία κάρτα βρίσκεται συνδεδεμένη αλλά δεν έχει ψηφίσει ο κάτοχος της κάρτας. Ρωτάω μήπως κάποιο μηχάνημα δεν λειτουργεί. Έχετε πατήσει όλοι τα πλήκτρα. Ανησυχώ λίγο γιατί έχουμε 44 κάρτες συνδεδεμένες και έχουν πατηθεί μόλις 43 κούμπια. Κάποιος λοιπόν μήπως σε κάποιον δεν ανάβει το φωτάκι. Κάποια κάρτα ίσως έχει βγει. Κλείνουμε λοιπόν την ψηφοφορία. 38 είναι υπέρ, ένας είναι δυσαρεστημένος και τέσσερις απήχαν. Περνάμε στην ψηφοφορία για τη δική μου έκθεση. Δεν είμαι σίγουρη ότι θα έπρεπε να βρίσκομαι στη θέση της Προέδρου. Έγινε από την Προεδρία εκ μέρου της ε, Επιτροπής για την ίσα ε, η τροπολογία 45 ε, συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά 51 votes open we have it's everybody voted votes ε, κλείνει η ψηφοφορία απορρίπτεται Προφορική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 11 υπέρ, κατά, εγκρίνεται 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική β, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά,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 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 28 υπέρ, 15 κατά, 60 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 16 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 17 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική C υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 62 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε Ψήφισαν όλοι ε, κλείνει η ψηφοφορία. Έχουμε μια ψηφοφορία υπερβολική, αλλά εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. 22 υπέρ, κατά, ε, αποχές, μπορούμε να ελέγξουμε την 22. Ελέγχουμε την 22. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται 28 υπέρ, 16 κατά. Ε, συμβαστική η ε υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά να το ελέγξουμε άρχεται η ψηφοφορία Ρέτζι 5 κλείνει η ψηφοφορία εγκρίνεται 31 υπέρ 11 κατά Ρέτζι 8 6 6 έκανε λάθος ο πρόεδρος 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές μπορούμε να την ελέγξουμε την 25 η ε, λίστα ψηφοφορία του εισηγητή είναι σύν αυτή τη στιγμή, μια αλλαγή τη τελευταία στιγμή. Έχουμε βάλει συν. 25 ε, υπέρ εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. Συμβεβαστική H υπέρ. Κατά. αποχέ εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 30, 31 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 33 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 35 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβιβαστική J υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ωραία λοιπόν ας ψηφίσουμε για ολόκληρο το κείμενο όπως τροποποιήθηκε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. 41 υπέρ, 1 κατά, δύο αποχές. Επαναλαμβάνουμε για το νομοθετικό ψήφισμα. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Ένας ΕΛΚ παραπάνω. Μπορεί κάποιος να προσυνδέσει. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. 39 υπέρ. 0 κατά, δύο αποχές. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και συζητητές και το προσωπικό που δούλεψε πολύ σκληρά στη γραμματεία. Ευχαριστούμε. Περνάμε τώρα, αν δεν κάνω λάθος... Είστε όλοι έτοιμοι για να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία για την έκθεση της Μαριαν Τάισεν για την κοινή ενοποιημένη εταιρική φορολογική βάση. Έχουμε μαζική ψηφοφορία για 14.59 υπέρ κατά αποχές συμβιβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σελίδα 3. Συμβιβαστική Β. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στη σελίδα 15. Συμβιβαστική C. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε στη σελίδα 18. Μαζικά μέχρι που, από τη σελίδα 18 είναι το μπλοκ που αφαιρεί το consolidation υπέρ κατά εδώ μιλάμε για τη σελίδα 18 είναι ένα ενοποιημένο μπλοκ ε, τροπολογίες 101 έως κάποια τροπολογία τη σελίδα 25 και μιλάμε εδώ για την αφαίρεση του όρου consolidation ενοποίηση, ενοποιημένη. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Απορρίπτεται μαζικά. Όλο αυτό θέλετε να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Εντάξει λοιπόν να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, είναι ένα σημαντικό σημείο, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Καλύτερα να είμαστε βέβαιοι. Ψήψαν όλοι, κλείνει η ψηφοφορία. Απορρίπτεται 39 κατά 12 υπέρ. Περνάμε στη σελίδα 25 τροπολογία. Είμαστε, είστε μαζί μου 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 147 8 και 9 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 50 και 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 152 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 153 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 154 υπέρ κατά αποχές εγκρι... απορρίπτεται 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 156 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ ΙΜΚΟ 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 158 υπέρ κατά αποχές Μπορούμε να το ελέγξουμε για την τροπολογία 158 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι πέρας ψηφοφορίας. 24 υπέρ εγκρίνεται, 24 έναντι 20. μαζευτείτε λίγο στην πρώτη σειρά. 159 ε, τροπολογία υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. ΙΜΚΟ 15 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 160 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική D υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα 189 υπέρ. Περιμένετε. Καταπίπτει. Περνάμε τώρα στην 2.10 έως 2.12 υπέρ. Η 189 καταπίπτει Ζαμπόλ. Οπότε είμαστε τώρα στην 2.10. 210 τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.28 και 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.45 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.56 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε τη 2.56 γιατί ήταν λίγα τα χέρια. Ψήφισαν όλοι, κλείνει ψηφοφορία 16, απορρίπτεται 16 υπέρ 28 κατά, 2.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 2.58 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.60 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.62 υπέρ κατά υπε, αποχές απορρίπτεται. 2.63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.64 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 2.67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 268 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 270 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ΙΜΚΟ 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 275 6, 7 και 8 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Τροπολογία 279 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 280 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 281 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 282 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 283 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 284 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 285 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται συμβιβαστική ε υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στην σελίδα 32, σελίδα 32, 340, 341 και 3... Ε, μάλιστα καταπίπτουν 343, ε, και 23, περνάμε σε 369, 379 γλωσσικά, 373 υπέρ κατά αποχές. Νομίζω ότι εγκρίνεται, το ελέγχουμε ηλεκτρονικά. 373 τροπολογία. ...373. Ψήφισαν όλοι. Κλείνει η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, 4 κατά. Κάποιοι άλλαξαν διάθεση. Εδώ 3,79, 80 και 81 υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 3,90 υπέρ, κατά, αποχές, ε, ε απορρίπτεται. 24, ε, υπέρ, κατά, αποχές, νομίζω εγκρίνεται. 391, 393 και 4 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ήμικο 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μεριάν. Ζητώ συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, η τροπολογία 4-3... 403 έως 408 έδωσα λανθασμένη ένδειξη ψηφοφορίας. Θα πρέπει να είναι αρνητική και θα σας πω γιατί αυτά, οι τροπολογίες αφορούν τις κατεξουσιοδότηση πράξης και την εντολή που δίνουμε στην Κομισιόν και οι τροπολογίες λέει ότι ουσιαστικά το Κοινοβούλιο πρέπει να εμπλέκεται κατά τον ίδιο τρόπο. Σημαίνει ότι μπορούμε να είμαστε υπευθύνοι για όλες τις ε, τεχνικές λεπτομέρειες και εγώ δεν πιστεύω ότι έχουμε τις ικανότητε για να κάνουμε κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει οργανική συμφωνία για αυτό το σκοπό. Είμαι λοιπόν κατά. Δεν το υποστηρίζω. Ε, εάν όμως η Επιτροπή έχει διαφορετική άποψη, ωστόσο εγώ ψηφίζω να, ε, προτείνω να ψηφίσουμε κατά. Θα πρέπει να είναι μείον και όχι συν. 403 406. All those in favour, against, abstentions, reject. Ε, απορρίπτεται 403 406, 407, 408 υπέρ. 407 και 408 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. 409-26 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 28 ΙΜΚΟ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4-2-1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 4-2-5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αυτό καταπίπτει 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 κατά πίπτη 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 23 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά α καταπίπτει συγγνώμη 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 υπέρ κατά αποχές. <coughs> Ελέγχουμε ηλεκτρονικά την 4. Τέλος, εγκρίνεται. 26 υπέρ 18 κατά. 5 κατά πίπτη, ΙΜΚΟ 5. 5 της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ΙΜΚΟ 6 είναι ίδια. 52 υπέρ. Α, καταπίπτει. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 καταπίπτει και η 62, όχι. Ψηφίζουμε την 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 63, 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 70 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 και 27 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μκο 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ήμκο 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική G υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91 καταπίπτει. Ήμκο 11, Ήμκο 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Η Μάριαν θέλει. Νομίζω ότι υπάρχει λάθος εδώ στον κατάλογο. Το 89 καταπίπτει γιατί ψηφίσαμε τη συμβαστική F. Η 89 ζητάει την αναθεώρηση μετά από τρία χρόνια. Ψηφίσαμε ήδη ότι θέλουμε μετά από πέντε χρόνια αναθεώρηση. Άρα η 91 καταπίπτει. 11 και 89. Α, εντάξει. Ωραία. Ίμκο 11, τροπολογία 89. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίσετε. Μη σταματάτε. Ίμκο 11 και τροπολογία 89. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Οκτώ υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το τροποποιημένο κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ένα ΕΛΚ επιπλέον. Δύο, δύο ΕΛΚ. Δύο ΕΛΚ παραπάνω ψήφισαν. Τέλος ψηφοφορίας. 35 υπέρ, 7 κατά μία εποχή. Το νομοθετικό ψήφισμα ψηφίζουμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 35-7-1. Συγχαρητήρια Μαριάννα. Μπράβο. yes. Yeah. Chair, in a spirit of transparency, I had promised the, rapport. Υποσχέθηκα στην ε, εισηγήτρια θα την καλέσω για δείπνο. Δεν ξέρω αν αυτό θα θεωρηθεί διαφθορά. Εν πάση περιπτώσει, θέλω όλοι να ξέρουν. Δέχομαι την πρόσκληση του Φιλίπ Δεύτερον. Θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω όλους, όλους τους συναδέλφους. Ήταν πολύ δύσκολο το θέμα, 400 τροπολογίες. Ξεκινήσαμε από πολύ διαφορετικές απόψεις, αλλά συζητήσαμε, βρήκαμε συμβιβασμό και πιστεύω πραγματικά ότι θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι στην Επιτροπή, να συνεχίσουμε την επεξεργασία του θέματος αυτού. Δεν είναι πάντα εύκολο να υπάρχει συμφωνία και ομοφωνία σε θέματα φορολογίας. Ευχαριστώ τους συγητές, ευχαριστώ τους κοιόδης, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος γιατί βλέπετε ότι υπάρχει μεγάλη πλειοψηφία και τώρα περνάμε στο επόμενο θέμα. Δύο λεπτά. Θα ήθελα εξ ονόματος της σοσιαλιστικής ομάδας να ευχαριστήσω την Μαριάν Τίσεν. Με ακούτε? Μαριάννα. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Κάτι που δεν είναι αγγλικά ακούγεται από το αγγλικό κανάλι. οκ. okay. Moi, je voulais juste remercier euh, Marianne Thyssen Θέλω να ευχαριστήσω την Μαριάν Τίσεν για την εξαιρετική της εργασία, για το ανοιχτό πνεύμα που έδειξε. Δεν ήταν εύκολο να φτάσουμε σε αυτήν την συμβαστική λύση. Πρόκειται για μια ευρεία συνένεση, η οποία πραγματικά ενισχύει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Okay, thank you very much. now moving Ευχαριστώ πολύ. Omnibus 2. Και υπάρχει και μία μικρή διαφορά εδώ σε σχέση με τον κατάλογο ψηφοφορίας στο τέλος, εν πάση περιπτώσει. Θα συνυπολογίσω όλους τις ψήφους. Uh, εν περιπτώσει, Φαντάζομαι όλοι όταν φτάσουμε στο σημείο αυτό, στο τέλος πληροφορίας, θα καταλάβετε. Τροπολογία 1 είναι τεχνική. Δεν ψηφίζουμε. 25 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική α υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ. 31. 27-31. 27-31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 32 αποσύρεται. 33 με 35. Μάλλον 33 με 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 315 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 383 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 403 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. 46 με 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική σι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Και 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική E, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 50, όχι. Συμβιβαστική F, υπέρ, κατά, αποχές, δεν βλέπω καλά. 56, 58 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 5, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. G, συμβαστική G, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64-65 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 339 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική γιώτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3-4-2 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικά ψηφίζουμε την 3-4-2 voted Τελειώσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 73 υπέρ και 74 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3-4-3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Απορρίπτεται, συγγνώμη, 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 3, 4, 5. Όχι, όχι. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 3, 4, 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική J και K υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα από 78 έως 80 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 371 καταπίπτει ή όχι. Όχι. Ψηφίζουμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Την ψηφίζουμε την 371. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να ελέγξουμε ηλεκτρονικά. 371. Ψηφίσατε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 375 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται ψηφίζουμε όμως ηλεκτρονικά δεν είδα ψηφίσατε όλοι τέλος της ψηφοφορίας η 375 απορρίπτεται 81 απορρίπτεται 81 και 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 με προφορική υποτροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 86. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 καταπίπτει. 373 καταπίπτει. 84 και 85 υπέρ. Και 87. Κατά αποχές εγκρίνονται. 88 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ο 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 91, 97. 91 με 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 377 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Όχι. 98 809 Εγκρίνεται, δεν βλέπω καλά. 88-109, συγγνώμη. Και περνάμε στην 378-379, υπέρ, κατά, αποχές. 380, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 381 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να ελέγξουμε όμως ηλεκτρονικά ...381, ψηφίσατε όλοι, τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 382 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική ε, προφορική υποτροπολογία υπέρ. Κάτι γίνεται. Ναι υπέρ, κατά, αποχές, δεν ξέρω ακριβώς, μάλλον εγκρίνεται. Συμβιβαστική, ποια συμβιβαστική είναι εδώ. Έμα, μη, που επίσης έχει προφορική υποτροπολογία. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Και τώρα μόνο η συμβαστική μη, εμ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. «135 μέχρι 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 407 υπέρ κατά όχι 407 στη σελίδα 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 153 μέχρι 157 υπέρ 153 έως 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική 1 νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 161 υπέρ μέχρι το 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική όμικρον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και 170 και 170 μέχρι την 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική π υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 422 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική R ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 και 189 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική S. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εκατόν μέχρι 200 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική ταφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 435 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 211 μέχρι 19 και 4.36 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβιβαστική W υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 230 μέχρι 236 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4-3-7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 2-3-7. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2-3-8. Μέχρι 2-5-5. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική. Χ. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 2 6 ε, συγγνώμη, με 2,70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τζούρι 1 καταπίπτει. Συμβιβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Z υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 279 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 280 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΑ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΑΒ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 282 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 472 υπέρ. 472 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 κατά πίπτη, 287 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 288 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 289 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 290 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 291 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 292 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 293 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 294 κατά πίπτη 295 το ίδιο 4 έχει αποσυρθεί 296 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται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 2-6-9 έχει εγκριθεί. 9, έχει εγκριθεί 300 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 11 υπέρ κατά αποχές 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 301 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 303 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Α, καταπίπτει 15. 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 305 καταπίπτει. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 306 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 306 Κάποιος από το ΕΛΚ έχει ψηφίσει δύο φορές. Ψηφίσατε όλοι. 19 υπέρ, 22 κατά. Απορρίπτεται. 18 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 307 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 308 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 309 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 310 310 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 310 310 310 310 310. 310. 310. Hang on, we got to confuse. Against. 300, 310, the rapporteur's list. Λοιπόν, υπάρχει ένα αρνητικό σήμα στον κατάλογο. Κυρία Πρόεδρε, το ερώτημα είναι τι ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το 309 γιατί το ΕΛΚ είναι υπέρ. Αν ψηφίζουμε το 3 310, το ΕΛΚ είναι κατά. Άρα πείτε μου, για ποιο ψηφίζουμε. Το 310 ψηφίζουμε. Κατά είναι ο εισηγητής και υπάρχει κάποιος από το ΕΛΚ που ψήφισε τουλάχιστον δύο φορές. Ωραία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Απορρίπτεται. 20 υπέρ, 23 κατά. 3-11 υπέρ κατά αποχές μάλλον απορρίπτεται αυτό ελέγχουμε εντάξει Μήπως δεν απορρίπτεται. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η 311. 312 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με σαφήνεια. Προφορική τροπολογία τελική σκέψη 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 313 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίζουμε το νέο κείμενο υπέρ κατά αποχές. Τέλος. 38 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Το νομοθετικό ψήφισμα, αρχή της ψηφοφορίας, ψηφίζουμε. Συνεχίστε να ψηφίζετε. Πάλι ένας από το ΕΛΚ έχει ψηφίσει δύο φορές. Τέλος της ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Yeah, okay. right. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Σας παρακαλώ, έχουμε και κάποια άλλα θέματα. Ο εισηγητής. Κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους τους κοιόδης εισηγητές. Ήταν όντως προκλητικό το θέμα, δύσκολο, τεχνικό και Πιστεύω ότι η συνεργασία υπήρξε πολύ επικοδομητική, το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ καλό. Ευχαριστώ όλους τους εισηγητές αλλά και σκιώδεις και όλους όσους συμμετείχαν. Περιμένετε, δεν τελειώσαμε ακόμη. Ο Σβέν θέλει να πει κάτι και μετά θα επανέλθω πάλι στον εισηγητή. Ο Σβέν. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους σκιώδεις εισηγητές και την πλειοψηφία για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Νομίζω ότι ήταν η ομόφωνη η συμφωνία που επιτύχαμε για τις συμβαστικές. Κάτι όμως έγινε κατά διάρκεια της διαδικασίας που μέχρι τώρα σε αυτήν την Επιτροπή δεν το είχα δει. Πρώτα απ' όλα, υπήρχε ισχυρή πλειοψηφία μεταξύ των σκιωδών εισηγητών για να εκφράσουμε μια ισχυρή θέση για το matching premium και όλα αυτά έγιναν παρά τα συνεισφορές που είχαμε κατά τη διάρκεια των ε, συναντήσεων που είχαμε και για την ε, ασφαλιστικά ταμεία στην Ευρώπη και την ρευστότητά τους ε, υιοθετήσαμε κάποιες θέσεις που ήταν πολύ καλές. Πρέπει να πω ότι ήταν ασύνηθες το ότι τα συμβιβαστικά κείμενα τα οποία είχαμε στο Κοινοβούλιο πηγαινόρχονταν μεταξύ ε, του κλάδου για τον οποίο ασχολούμεθα και ημών σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης. Αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε, διότι διέρευσαν κάποια κομμάτια στον τύπο πριν εμείς να μπορέσουμε οι σκιώδεις εισηγητέ να δούμε κάτι. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσάψω στον εισηγητή, ο οποίος ήταν πάντα πάρα πολύ σωστός, αλλά όλα αυτά τα θέματα θα πρέπει να τα συζητήσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών και ελπίζω ότι δεν θα γίνει πάρα πολύ χειρότερη κατάσταση από ότι είναι, διότι σε θέματα ε, ρευστότητας εμείς έχουμε κάνει κάποια πράγματα εδώ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί μεταξύ μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για το εξαιρετικό του έργο. Έχουμε εδώ μια πολύ ισορροπημένη μέτριων με την οποία όλοι συμφωνούμε. Για να είμαι ειλικρινής, ε, κοιτώντα ε, τις επιπλοκές που είχαμε στο, επίπεδο, στο πρώτο επίπεδο του κειμένου που παρουσιάστηκε για την νομική αξιολόγηση εδώ, ε, μιλάμε και για πολιτικούς ακροβατισμούς εκείνη την εποχή. Πιστεύω λοιπόν ότι είχε επιτευχθεί εξαιρετική ισορροπία. Ακούω κάποια σχόλια από κάποια άλλα μέλη του Κοινοβουλίου, αλλά ας είμαστε ειλικρινεί. Από την εμπειρία μου εδώ και 20 χρόνια σε αυτό τον οίκο πολλά συμβαίνουν. Είμαστε μια δημοκρατικά, ένα δημοκρατικά εκλεγμένο κοινοβουλίο. Χρειάζεται ανάλυση στην Επιτροπή. Η ομάδα εργασία ε, δεν είχε καταφέρει να επιτύχει την ε, ισορροπία που βλέπουμε τώρα. Υπήρχε μεγάλη διχογνωμία. Εγώ δεν είμαι πεπισμένο, ωστόσο, ότι έχουμε βρει όλε τι απαντήσει που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά χρειάζεται να σημειώσουμε πρόοδο και χαίρομαι ιδιαίτερα που έχουμε καταφέρει να επιτύχουμε αυτό το συμβιβασμό σήμερα. Ευχαριστούμε λοιπόν και τον εισηγητή και του Σκιώδη. Ευχαριστώ. Θα πρέπει να έχουμε το νου ότι πολλές φορές τον επανέρχονται κάποιες εκθέσει στις ομάδες. αλλάζουν τα πράγματα διαφορετικά από το πριν. Και πολλές φορές είναι δύσκολο πάντα να ξέρουμε τι θα συμβεί και πότε και προς τα ποια κατεύθυνση. Έγινε η ψηφοφορία, είχαμε μεγάλη πλειοψηφία υπέρ και θα ήθελα να μου πει τώρα ο εισηγητής ε, εάν προτίθεται να κάνει διαπραγματεύσεις ε, σε επίπεδο των τριών οργάνων για να μπορέσει να επιτευχθεί η ε, συμφωνία σύμφωνα βεβαίως με την συνηθισμένη διαδικασία και ο συνήθως οι σκιώδεις εισηγητές, ο εισηγητής και η πρόεδρος θα συμμετέχουν σε όλη αυτή την δικασία όπως ξέρουμε. Αλλά ας δώσω το λόγο στον εισηγητή να μας τα εξηγήσει αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτό που είναι σημαντικό είναι από εδώ και πέρα οι συζητήσεις που θα λάβουν χώρα μεταξύ Επιτροπής και Συμβουλίου και ημών και βεβαίως να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκινήσαμε. Πολύ καλά. Μπορώ και εγώ προ... Σωρινά να σε επιβεβαιώσω ότι η πρώτη συνάντηση σε επίπεδο τριών οργάνων θα γίνει 11 Απριλίου. Επίση, θα ήθελα να πω ότι 29 11 θα γίνει η ψηφοφορία η τελευταία, αφού έχει γίνει εκ των προτέρων η πρώτη συνάντηση και η πρώτη ψηφοφορία ε, σε επίπεδο πρώτης ανάγνωσης. Όπως ξέρετε, η ομάδα διαπραγματευτική θα είναι η συνήθις. Επίσης, θα ήθελα να σας επενδυμίσω ότι πρέπει να επανέλθουμε στις 3, διότι έχουμε ανταλλαγή απόψεων με τον ε, Επίτροπο Μπαρνιέ. Ο Ζων Πολ θέλει κάτι να πει. Δεδομένου το τι έγινε στις τελευταίες συνεδριάσεις, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι όπως μας υποδείξατε, η εντολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι η έκθεση. Και ο διάλογος μεταξύ των τριών οργάνων δεν θα πρέπει να αποτελέσει πρόσχημα για να τεθεί ή ένα αμφιβόλο ότι ψηφίστηκε εδώ από την Επιτροπή ή να προσπαθήσουν να επικρατήσουν οι απόψεις με ψηφίες. Το λέγω γιατί έχει ξαναγίνει. Ε, λοιπόν, θα ήθελα εσείς να κάνετε ό,τι μπορείτε για να τηρηθεί η εντολή και έτσι ως έχει και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το ίδιο θα πράξει και ο εισηγητής. Ευχαριστώ. Η Αστριντ. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία ελέγχθησαν τώρα. Δεν καταλαβαίνω όμως τι είπε ο κύριος Γκίγκον. Διότι πολλές φορές με τους φιλελεύθερους και τους σοσιαλιστές κάνει διάφορους συμβιβασμούς ε, πίσω από την πλάτη μας και τώρα εκνευρίζεται. Τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά. be Είναι πολλές φορές επώδυνη η δημοκρατία, λένε ό,τι καλύτερο έχουμε. Γεια σας, ραντεβού και πάλι στις τρεις.